Αρχίζουμε τις ψηφοφορίες. Μπράβο. Προβλέπει την ψηφοφορία σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία επί της έκθεσης του κυρίου Καρίμ σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την αναγνώριση της πατρίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο. Τη θέτω σε ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Roll call vote. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση καρύμ σχετικά με την προσέγγιση νομοθεσιών κρατών μελών των αναφερομένων στις μονάδες μετρήσεως με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Καρύμ σχετικά με το αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και την διάταξη εξατμίσεως των μηχανοκίνητων οχημάτων. Με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα σοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Καρύμ σχετικά με τη δομή προστασία σε περίπτωση ανατροπής τοποθετημένη στο εμπρόστιο μέρος των τροχοφόρων γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο με ονομαστική κλίση άρκετη η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Καρύμ. What's the problem? Your machine is not working. Okay, we'll send someone there. 463, I think, yes. Έκθεση Καρύμ σχετικά με την εγκατάσταση, τοποθέτηση, λειτουργία, αναγνώριση οργάνων χειρισμού των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με τροχούς. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Καρύμ σχετικά με την πέδηση των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας οφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Καρύμ σχετικά με το διαθέσιμο χώρο χειρισμού, την ευχέρεια πρόσβαση στη θέση οδήγηση καθώ και τι θύρε και τα παράθυρα των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχού. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση Καρύμ σχετικά με τη δομή προστασία σε περίπτωση ανατροπή τοποθετημένη στο οπίστιο μέρο τροχοφόρων γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση Καρύμ σχετικά με τη διάρθρωση και του συντελεστέ του ειδικού φόρου κατανάλωση που εφαρμόζονται στα βιομηχανικά καπνά. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα οφορίας, Εγκρίνεται. Ε, έκθεση Καρίμ. Σχετικά με την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα οφορίας, Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Καρίμ. έκθεση Manders σχετικά με τις ονομασίες των υφανσίμων ινών και τη συναφή επισήμαση και σήμανση σύνθεση ινών των κλωστοβιωτικών προϊόντων. The rapporteur wants the floor. Mr. Manders. Ο εισηγητής θέλει το λόγο. Ο κύριος Μάντερς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει εδώ μια κοινή δήλωση στην οποία συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο. Ο... Η αρμόδια υπουργό, κυρία Γιώργιου, Γιώργη, ε, μου είπε να την αναγνώσω εγώ γιατί δυστυχώ δεν έχει φωνή. Λέει τα εξή στα αγγλικά. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αναγνωρίζουμε τη σημασία του να υπάρχει σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών, ιδίως όταν τα προϊόντα τη χάνουν εμπορία χωρί ε, συγκεκριμένη αναφορά προέλευσης. Για να προστατεύσουμε λοιπόν τους καταναλωτές κατά παραπλανητικών πληροφοριών, η χρήση των νέων τεχνολογιών και η ηλεκτρονική ετικετοθεσία, μεταξύ των οποίων και τη χρήση ε, ραδιοσυχνοτικών ετικετών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λαφθεί υπόψη η τεχνολογική αλλαγή. Το Συμβούλιο λοιπόν και το Κοινοβούλιο καλούν την Κομισιόν όταν συντάξει μια έκθεση βαστού του 24 24α να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών για τις νέες ανάγκες τοθεσίες, ιδίως για την ανεχνευσιμότητα των κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων και ελπίζω τώρα ότι το Συμβούλιο θα συμφωνήσει. Πάμε τώρα στην ψηφοφορία. Τροπολογία 35. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει το μπλοκ 2 και η πρόταση υιοθετείται από την Ολομέλεια. Συγχαρητήρια στον κύριο Μάντερς. Έκθεση Μορέιρα. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. I'm sorry. There's no amendment 14. Υπάρχει μια προφορική τροποποίηση στο, στην τροπολογία 14. Έχετε το λόγο κύριε Μουρέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια προφορική τροπολογία στη δική μου έγγραφη τροπολογία 14 και λέει τα εξής η τροπολογία. Εκεί που λέει χώρες προτείνω να πούμε χώρες και εδάφη. Ο στόχος αυτής της προφορικής τροποποίησης είναι προφανής. Για να ευθυγραμμιστεί η διατύπωση αυτής της παραγράφου με τον τίτλο του ίδιου αυτού του κανονισμού. Γιατί ο τίτλος λέει τα εξής, παραθέτω, έκτακτα εμπορικά μέτρα για χώρες αλλά και για εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με, με την ε, διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς αυτή την ε, αλλαγή θα υπήρχε μια διαφορά μεταξύ του περιεχομένου του κανονισμού και του τίτλου. Γι' αυτό ζητώ την υποστήριξή σας για να γυρθεί αυτή η τροπολογία. Σε αυτή την προφορική τροπολογία, any objections? Για to stand up if you have an objection. Okay, uh, επομένως, they're not 40, I'm sorry. Επομένως, ε, we vote on uh, amendment 14 with the oral amendment. Ψηφίσουμε την τροπολογία 14 με την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Let's check. 14. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη 14. Άρχεται. Πέρα της εγκρίνεται. τροπολογία 15, 15. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. 18. You want to check on 18? I said εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο στην 18. Ε, Είπα ότι εγκρίνεται, αλλά κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Θα σας πω τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Επειδή μπορείτε να νομίζετε ότι χρειαζόμαι βοήθεια σε αυτή την ε, ψηφοφορία, με βοηθάτε. Όποιο θέλει έλεγχο θα πρέπει να στέκεται όρθιο, θα ελέγχουμε. Αν είχα δίκιο θα πρέπει να πει στα ελληνικά εγκρίνεται κύριε Πρόεδρε ή απορρίπτεται κύριε Πρόεδρε. Εντάξει. Τροπολογίες 8 με 10. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Έχει withdrawn. Με συγχωρείτε. 22 υπέρ κατά uh, I'm confused check 22 έλεγχος για την 22 believe it πέρας οφορίας εγκρίνεται 12 <laughs> ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 ε, σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, η πρόταση όπως έχει τροποποιηθεί, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, ο κύριος Μορέιρα θα ήθελε ε, το λόγο. Κύριε Μορέιρα. You have asked for the floor, I understand. Θέλετε το λόγο κύριε Μουρέιρα. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ζητήσω αναβολή της, ε, του νομοθετικού ψηφίσματος. Η Επιτροπή έχει κάτι να πει από αυτού. Does the Commission have something to say on this? The Commission welcomes... Uh, Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόταση του κύριου Ευρωβουλευτή, διότι μας δίνει χρόνο για να εξετάσουμε καλύτερα τις τροπολογίες και υπάρχει και χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να, ε, τον οποίο μπορούν να εκμεταλλευτούν για να καταλήξουμε σε ε, ψηφοφορία. Επομένως υπάρχει πρόταση για να επιστρέψει στην Επιτροπή. Αποχές εγκρίνεται. Επιστρέφει η πρόταση στην Επιτροπή. Έκθεση Χόκμαρκ σχετικά με την καθιέρωση του πρώτου προγράμματος πολιτικής για, τα, για, το ραδιοφάσμα. Ε, το πρώτο μπλοκ τροπολογιών από την Επιτροπή ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 σε δύο μέρη. Με ονομαστική κλίση. Πρώτο μέρος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 69 σε δύο μέρη με ονομαστική κλίση. Πρώτο μέρος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 90. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, η ψήφος επί της προτάσεως όπως έχει αναθεωρηθεί ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με ονομαστική κλίση το ψήφισμα άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Χόκμαρκ Περνάμε τώρα στην έκθεση Κασίνη σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνέχεια της δημιουργίας κοινού μητρώου διαφάνειας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Dear colleagues, I have a statement to read. να σας διαβάσω μία δήλωση. Η έκθεση Καζίνη για τη διαθεσμική συμφωνία σε σχέση με ένα κοινό μητρώο διαφάνειας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κομισιόν εκπροσωπεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για να ρυθμιστούν οι σχέσεις αυτών των φορέων με εξωτερικές οντότητες. Πριν ψηφιστεί αυτή η έκθεση θέλω να υπογραμμίσω ότι οι συνεχιζόμενες εργασίες της ομάδας εργασίας για τον κώδικα Συμπεριφάσεις των βουλευτών και τα εξωτερικά συμφέροντα δεν έχουν σαν στόχο να ανατρέψουν την ουσία της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί με την Κομισιόν και το περιεχόμενο της έκθεσης Καζίνη. Έχουν σαν στόχο να συμπληρώσουν το πλαίσιο αυτό προσθέτοντας νέες πτυχές και ιδίω να ενισχύσουν του κανόνε που εφαρμόζονται σε σχέση με την πρόσβαση των ομάδων πιέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στου χώρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αμήν, λέει ο πρόεδρο. Εντάξει, όλοι έτοιμοι. Τροπολογίες 1 με 13 από κοινού. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, ψήφος, τελική ψήφος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, έκθεση Κασίνη σχετικά με, τροποποίηση, ε, σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής σχετικά με το κοινόμητρο διαφάνειας. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος <laughs> I'm, going to pretend I didn't hear this. Θα κάνω ότι δεν το άκουσα αυτό. Σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ Κατά. Αποχές. Check. Amendment 3. Έλεγχος τροπολογία 3. Πέρας οφορίας. Α, οκ. <laughs> Οκ, οκ. Uh, that's fine. So that's εγκρίνεται then. Uh, final, uh, well, uh, paragraph one. Paragraph nine. But wasn't this approved? Was no, rejected. Okay. Original text of paragraph 9. Αρχικό κείμενο στην παράγραφο 9. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψήφος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Κασίνη. Έκθεση Fox σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τροπολογία 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 1 με 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τελική ψήφος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Φόξ. Τέσσερι προτάσει ψηφίσματο σχετικά με την κατάσταση πραγμάτων στι διαπραγματεύσει για Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδία. Τροπολογία 7. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 σε δύο μέρη με ονομαστική κλίση πρώτο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. We go to the second part. Δεύτερο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας οφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέραση οφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 σε δύο μέρη με ονομαστική κλίση πρώτο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11 σε δύο μέρη με ονομαστική κλίση. Πρώτο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρο... Who said this? Who said this? Who said this? I want... Ποιος το είπε? Was that you, Mr. Wieland? Εσείς κύριε Βίλαντ. Εντάξει κύριε Αντιπρόεδρε. What did I say? Did I say εγκρίνεται or απορρίπτεται? I said εγκρίνεται. Okay. Now, any one of you, this is not an important issue you want to... Είναι σημαντικό θέμα. Αν θέλετε να αλλάξετε, να αλλάξετε την ψήφα σα και να εγκρίνετε, αυτό είναι ευκαιρία σα. Ηλεκτρονικός έλεγχος, στην τροπολογία 4. Πέρα της ψηφοφορίας. I want you to stand up. Εγκρίνεται, Mr. Πρόεδρε. Thank you. Σηκωθείτε και πείτε εγκρίνεται, κύριε Πρόεδρε. Α, ευχαριστώ. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Με, ονομαστη... <laughs> Με ονομαστική κλίση. Ε, η τελική ψήφος. αρκετή ψηφοφορία. Πέρα της οφορίας εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στους συντάκτες. Τώρα, ε, η μερίσια διάταξη προβλέπει ψηφοφορία τέσσερις προτάσεις ψηφίσματος σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας. Τροπολογία 1 σε δύο μέρη. Α. We will start with an oral amendment by Mr. to paragraph 2 με Προφορική τροπολογία του κυρίου Βαλέσα στην παράγραφο 2. Κύριε Βαλέσα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, για τη συγκεκριμένη τροπολογία το ΕΛΚ ζητά να διαγράψουμε τον όρο strongly στην παράγραφο 2. Ελπίζω να μην υπάρχουν ενστάσεις. Ευχαριστώ. Υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτή την προφορική τροπολογία. Όχι. Άρα ψηφίζουμε την παράγραφο 2 με την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψήφος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η μερίστη διάταξη προβλέπει ψηφοφορία από τις έκθεση του κυρίου Αρσένη σχετικά με την προστασία και την προετοιμασία των δασών εν ώψη κλιματική αλλαγή. Παράγραφος 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 25 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται check second part of 25 ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα του 25 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται παράγραφος 36 σε δύο μέρη πρώτο μέρος ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δεύτερο μέρος, υπέρ. Α, κύριε Σένη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορώ βέβαια να πω σε κανέναν να καταψηφίσει την απαγόρευση για τις καμές σε περιοχές οι οποίες είχαν ε, ε, καεί από φωτιές ε, για παράνομους σκοπούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για όλες τις χώρες Ευρώπης. Και αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 36 δεύτερο τμήμα και παράγραφο 37 προσπαθεί να διασφαλίσει την νομιμότητα και να καταπολέσουμε τις παρανόμες δραστηριότητες ε, στα δάση στην ε, Ευρώπη. Ζητώ λοιπόν να υπερψηφίσετε όλοι το 36β και την παράγραφο 37. Ε, οπότε σε ονομαστική κλίση θα βάλουμε το δεύτερο μέρος της 36 και την Παράγραφο 37. Okay. Second, second part of 36 by roll call vote. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 37 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της φοβορίας. Εγκρίνεται. Ε, παράγραφος 59. Ποιοι είναι υπέρ. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71 σε δύο μέρη. Πρώτο Πρώτο υπέρ. Κατά. Κατά. εγκρίνεται. Δεύτερο Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 σε τέσσερα μέρη. Πρώτο μέρο υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρο υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Check second part of 72. Δεύτερο τμήμα Πέρας οφορία. Απορρίπτεται. Τρίτο μέρος. Υπέρ. Third part. Τρίτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Check. Check the third part. Έλεγχος του τρίτου μέρους. Ε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τέταρτο μέρος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, recital H σε τρία μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται I'll check the second part. Θα ελέγξω το δεύτερο τμήμα. Πέρας οφορία. Oh, come on. You did not raise your hands right. Ε, παιδιά, δεν σηκώσατε τα χέρια κανονικά. third part. Τρίτο μέρος, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψήφος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Αρσένη. Έκθεση Αλμπερτίνη σχετικά με τι κύριε πτυχέ και τι βασικέ επιλογέ κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια για το 2009. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 2 Ποιος θέλει το λόγο. Ορίστε κύριε Χίχεστερ. Πρόεδρε, βλέπω ότι διασκεδάζετε εδώ με τον ανορθόδοξο τρόπο που διευθύνεται τη συζήτηση και με τα αστιάκια σας, αλλά εγώ προτείνω να είστε λίγο πιο αργός για να προλαβαίνουν και οι διερμηνείς. Τότε μπορούμε να ψηφίζουμε καλύτερα. Είστε λίγο γρήγορος και ως αποτέλεσμα καθυστερούμε. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Χίχεστερ. Κατά αυτό που είπατε καταλαβαίνω ότι εγκρίνετε τους ανορθόδοξους τρόπους μου. Okay. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είκοσι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές ε, check 3 έλεγχος 3 πέρας σοφορίας απορρίπτεται ε, ο κύριος Αλμπερτίνη έχει μια προφορική τροπολογία στο αρχικό κείμενο της παραγράφου 33 Κύριε Αλμπερτίνη, έχετε το λόγο. Περιτώ να το παραθέσω. Αναφέρεται στην ε, δήλωση ψήφου. Ξεκινάει με το Welcomes και ολοκληρώνεται με το Manner. Μπορείτε να το διαβάσετε στο κείμενο. Υπάρχει καμία αντίρρηση σε αυτή την τροπολογία? Όχι. Επομένως ψηφίζουμε παράγραφο 33 με την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ? Ποιοι είναι κατά? εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο παραγράφου 38 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος με ονομαστική κλίση. Άρκετη ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία στην τροπολογία 7 από τον κύριο Αλβερτίνη. 7. 7. That's correct. Προφορική τροπολογία στην τροπολογία 7 από τον κύριο Αλμπερτίνη. Mr. Αλμπερτίνη, Κύριε Αλμπερτίνη, έχετε το λόγο. Ναι, και σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνεται στον κατάλογο ψηφοφοριών το κείμενο. Ένα σχόλιο μόνο αφορά την ε, διαμαρτυρία για τις καταδίκες των ε, διαδηλωτών στο Μπαχρέιν και την λογοκρισία επί του συγκεκριμένου θέματος. No, that's, uh, Κύριε Αλμπερτίνη, μιλάω για την προφορική τροπολογία στην ε, τροπολογία 7 μετά από την παράγραφο 45. Α, συγγνώμη, διάβασα λάθος κείμενο, λέει ο κύριος Αλμπερτίνη. Έχουμε αφαιρέσει τον όρο Μακεδονία γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες ευαισθησίες νομίζω και του Προέδρου σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει μόνο λοιπόν πλέον πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και δεν αναφέρεται το όρος Μακεδονία. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν παράγραφο 7 με την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. I'm sorry. Ποιοι είναι υπέρ. Εντάξει, έχουμε 40, άρα απορρίπτεται η προφορική τροπολογία και προχωράμε στην ψήφο επί της τροπολογίας 7 χωρίς την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας 7. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Οκτώ. υπέρ κατά αποχές check 8 άρχεται η ψηφοφορία πέρα ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 9 ποιοι είναι υπέρ Ποιοι είναι κατά. Ε, the e please raise your hands. παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 11. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 uh, και 24 καταπίπτουν 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται yes I have to echo Mr. Chichester's earlier intervention. In Grinita, I'm not aware that. Οι διερμηνεί λένε να πούμε όχι, να πούμε κατά, προτού ε, καθυστερημένα. Παρακαλώ, εάν θέλετε να μιλάτε ελληνικά, να μιλάτε πιο αργά. Μα απαιτείται να γνωρίζουν ελληνικά οι ευρωβουλευτές. Now listen. Μπορώ να τα κάνω και πολύ αργά όλα αυτά, αλλά... Αλλά δεν να μην αλλάζω τον τρόπο μου κάθε φορά. Λοιπόν, όπως ξέρετε όλοι οι διερμηνείς έχουν μπροστά τους τον κατάλογο ψηφοφορίας. Αν δεν τον έχουν να τον πάρουν. Και επομένως δεν αλλάζει το γρήγορο ή το αργό οι διερμηνείς έχουν μπροστά τους τον κατάλογο. Θα προσπαθήσω πάντως να είμαι λίγο πιο αργός, αν αυτό βελτιώσει τα πράγματα, δεν ξέρω. Τέσσερα. Yes, Mr. Yes, Mr. Dartmouth, you have the floor. Ορίστε, έχετε το λόγο. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Μιλάτε πολύ καλά αγγλικά και το έχετε δείξει. Αλλά γιατί επιμένετε εδώ πέρα να κάνετε αυτήν την παντομήμα. Τροπολογία 14. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 85 σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Mr. Albertini, you have the floor. I'm sorry. Κύριε Αλμπερτίνη, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη, δεν θα ήθελα να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι δεν ψηφίσαμε την προφορική τροπολογία στην παράγραφο 68. Αν δεν κάνω λάθος λοιπόν δεν έχουμε ψηφίσει την προφορική τροπολογία που είχα αναφέρει προηγουμένως για την καταδίγωση της ε, στάσης της κυβέρνησης του Μπαχρέιν. Πρέπει να την ψηφίσουμε λοιπόν. Η απάντηση σε αυτό κύριε Αλμπερτίνη είναι ε, υιοθετήσαμε τις τροπολογίες 13 ε, και 18 και η παράγραφος λοιπόν ε, στην οποία είχατε την προφορική τροπολογία κατέπεσε. Πέντε σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο μέρος με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τελική ψήφο. Ποιοι είναι υπέρ. Με συγχωρείτε. What? Mr. Mr. Goebbels, you have the floor. Yes, uh, Mr. President. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να υποστηρίξω τον κύριο Αλμπερτίνη, γιατί νομίζω ότι μπορούμε, θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε την προφορική του τροποποίηση ως προσθήκη στην παραγραφό που αναφέρεται. Θα ήταν θετικό να μπορέσουμε να καταδικάσουμε αυτά που γίνονται στο Μπαχρέιν, ιδίως τις θανατικές ποινέ εκεί. Κύριε Σφόμποντα και εγώ θέλω να το υποστηρίξω αυτό γιατί μάλλον ήταν σφάλμα στον κατάλογο ψηφοφορίας είτε στις ε, στάσεις μας στην ψηφοφορία. Είναι τόσο μεγάλη ομοφωνία που είναι παράξενο να μην υποστηρίξουμε τον κύριο Αλμπερτίνη και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι με την πρόταση να ψηφίσουμε αυτό το σημείο σαν πρόσθετο. Um, I think that's uh, fair. Εντάξει, σωστό είναι αυτό. Την ε, προφορική τροπολογία που μας παρουσίασε πριν ο κύριος Αλμπερτίνη ε, ως επιπρόσθετη ε, στην παράγραφο 68 ως έχει τροποποιηθεί από τις άλλες τροπολογίες. Ε, υπάρχει αντίρρηση στην τροπολογική τροπολογία. First of all, is there an objection to the oral amendment? Αντίρρηση στην προφορική τροπολογία. Είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τελική ψήφο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Αλμπερτίνη. Έκθεση Γκολτιέρη σχετικά με την ανάπτυξη της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας μετά την έναρξη ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 13, 20, 27, 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τέσσερα. με ονομαστική κλίση τροπολογία τρία. raise your hands υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία Πέρα ψηφοφορίας Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 7 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ε, με συγχωρείτε για να δούμε. Απορρίπτεται. 8 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 16. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15, 21, 28 και 30 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Υπάρχει μία... Is there No, no, the original text and amendment again. Okay, so we won't do the original text now. No, okay. 17. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Okay. Η τροπολογία 18 έχει αποσυρθεί και υπάρχει μία... Hold on a second everyone. Hold on a second. Μια στιγμή, μια στιγμή. Πρική τροπολογία στην παράγραφο 87 από τον κύριο Γκολτιέρη. Mr. Lisek, you had the previous oral amendment. You have the floor. Zgłaszałem Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα τραγικά γεγονότα της Λιβύης μας οδηγούν στο να πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια προσθήκη στην τρίτη σειρά μετά από την επιτόπια ανάπτυξη δυνάμεων θα θέλαμε να μιλήσουμε και για το εξή. Να δώσουμε άμεση ανθρωπιστική υποστήριξη για τη Μισουράτα και άλλα κέντρα του πληθυσμού, ιδίω από ναυτικέ δυνάμει και ανησυχούμε ιδιαίτερα για τον αυξανόμενο αριθμό θυμάτων τη σύγκρουση στη Λιβύη και τη χρήση βία από το καθεστώ Καντάφη. Κύριε Λίσεκ, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Έχει εκπέσει γιατί έχουμε εγκρίνει τις τροπολογίες για την παράγραφο 71. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να την ψηφίσουμε έχει τροποποιηθεί η τροπολογία από τις προηγούμενες τροπολογίες που ενεκρίθησαν. Εντάξει. Μια προφορική τροπολογία στην παράγραφο 87. Κύριε Κουαλτιέρη, έχετε το λόγο. Okay. Λένε το εξής οι προφορικές τροπολογίες ή μάλλον το πρωτότυπο λέει αναγνωρίζει ότι το ΝΑΤΟ είναι η βάση, το θεμέλιο της συλλογική ασφάλειας των μελών του. Και εδώ είναι η προσθήκη. Και πέραν αυτών, και πέραν αυτών. Όχι. Άρα ψηφίζουμε την παράγραφο 87 με την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Είχαμε ξεπεράσει την 12 νομίζω λένε ορισμένοι. Για το ξαναδούμε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οκ. Τελική ψήφος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Κουαλτιέρη. Αγαπητοί συνάδελφοι. Yes, please. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω ένα διαδικαστικό για την επόμενη έκθεση. Μονιές Διακούιζα, αν το πρόφερα σωστά. Ζήτησα αναφορά στο 161 για την τροπολογία 25 ένα συνάδελφο ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία γιατί θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και το είχατε εγκρίνει. Αλλά οι κανονισμοί προβλέπουν να ζητάτε πρώτα έγκριση από όλο το κοινοβούλιο. Αυτές είναι οι ανορθόδοξες μέθοδοι. Ζητώ λοιπόν και εγώ για μία ρήτρα που είναι ιδιαίτερα σημαντική για μένα να γίνει ονομαστική ψηφοφορία για όλες τις τροπολογίες της έκθεσης αυτής όπως δεχτήκατε και προηγουμένως για τον κύριο. Συνάδελφοι, η χορήγηση μία δίας για ονομαστική ψηφοφορία είναι κατά τον κανονισμό δικαιοδοσία του Προεδρεύοντος μπορεί να τη δεχτεί αν δεν διαταράσσεται η σύνοδος ή αλλιώς μπορεί να ρωτήσει το, την αίθουσα. Δεν υπάρχει όμως σαφής κανόνας, να το ξέρετε, για να μην δημιουργηθεί εδώ ψευτοπροηγούμενο. Υπό τις παρούσες συνθήκες λοιπόν, κύριε Σούλτς, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Να δεχτώ το αίτημά σας αυτή τη φορά αλλά παρακαλώ τους συναδέλφους να μην κάνουν κατάχρηση αυτών των δυνατοτήτων αλλιώς ο Προεδρεύων κάθε φορά θα ρωτάει και θα υπάρχει, υπάρχουν διαφορές και διχογνωμίες χωρίς να χρειάζονται λοιπόν. Αν επιμένετε να γίνουν όλες ονομαστικά, ορίστε. Με ονομαστική κλίση άρχεται προσφορία. Εγκρίνεται. Τέσσερα με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ένα με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πέντε με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, παράγραφος 20 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 26 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 31 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 32 σε δύο μέρη με ονομασία κλίση πρώτο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας εγκρίνεται 38 σε δύο μέρη πρώτο μέρος άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται δεύτερο μέρος άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 2 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τελική ψήφος με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ και συνάδελφοι. Και τώρα ακολουθούν οι αιτιολογήσεις ψήφου. Do we have Yeah.